Um, I will speak in uh, Portuguese. Um, boa tarde a todos. Vamos agora dar início. Uh, καλησπέρα σε όλους. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν το workshop ε, που διοργανώνεται λόγω και τις ε, ημέρες για την γυναίκα της Υπέθρου, την αγρότησα γυναίκα δηλαδή, που εορτάστηκε για πρώτη φορά το 2008 και με βάση το ψήφισμα των ΗΠΑ ναι, 62-136 που αναγνωρίζει ακριβώς το σημαντικό ρόλο της αγροτικής γυναίκας συμπεριλαμβανομένων των αυτόχων γυναικών στην αγροτική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της υπαίθρου στη βελτίωση της εμπιστητικής ασφάλειας και στην εξάλληψη της ε, ένδυας στις αγροτικές περιοχές. Έτσι λοιπόν καλέσαμε από την πλευρά της ε, Επιτροπής μας δύο επιρρογνώμονες οι οποίες ε, θα μας ε, κάνουν δύο παρουσιάσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πώς μπορεί να συμβάλλει στην κατάσταση των γυναικών στην Ήπειρο, στις αγροτικές περιοχές ή η κοινή γεωργική πολιτική. Επίσης θα συζητήσουμε ειδικότερα το ζήτημα του πώς ποιος είναι ο αντίκτυπος των ρόλων των γυναικών στις αγροτικές περιοχές σε ό,τι αφορά την απασχόληση και σε ό,τι αφορά και την εξορρόπηση ή την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά την απασχόληση σε αυτόν τον τομέα και κατά συνέπεια η ισότιμη πρόσβαση των δύο φύλων στις ίδιες ευκαιρίες στον αγροτικό τομέα. Άρα λοιπόν, οι ε, ε, πολιτικές των ε, κοινές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα σχετικά ταμεία θα πρέπει να αναλυθούν ως προς αυτή τη διάσταση. Ε, ε, προτού λοιπόν δώσω το λόγο στους δύο μελετές μας, θα δώσω το λόγο στην κυρία Νόης, ώστε να μας κάνει μια μικρή εισαγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Πετήρ καλώς εκείνη ήταν που πρότεινε την διοργάνωση της σημερινής συνεδρίας. Εσείς που έρχεστε από μια ε, αγροτική περιοχή και εγώ που έρχομαι από αγροτική περιοχή, οπότε ε, χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα σήμερα να κάνω αυτή την εισαγωγή σήμερα, αλλά σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά που διοργανώσατε τη σημερινή, το σημερινό αυτό workshop. Όταν μιλάμε λοιπόν για αγροτικές περιοχές, δεν μιλάμε για μια ενιαία αγροτική περιοχή, μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιμέρους, επιμέρους περιοχών, οπότε ε, ε δεν θα πρέπει να κάνουμε μια τέτοια διαφοροποίηση γενική μεταξύ μεταξύ δηλαδή της γυναίκας στην ε, αρχιστική περιοχή και τη γυναίκα στην ε, αγροτική περιοχή γιατί και οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μπορεί να βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις και η θέση τους δηλαδή μέσα στην αγροτική ε, περιοχή είναι διαφορετική μέσα στα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια οι αγροτικές περιοχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή πριν από 50 χρόνια οι περισσότερες γυναίκες στις αγροτικές περιοχές απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας. Αυτό όμως έχει αλλάξει σήμερα. Υπάρχουν νέα επαγγέλματα στις, ε, στις, στις ε, περιοχές της Υπέθρου, αλλά και σε κάποιες άλλες όχι. Και αυτό θα το συζητήσουμε και σήμερα. Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν για πολλούς ανθρώπους την Κυριακή έναν προορισμό εκδρομής. Θέλει να πάει κανείς εκεί δηλαδή για λόγους ψυχαγωγίας. Αλλά ε, τι συμβαίνει συμβαίνει με τις γυναίκες εκείνες οι οποίες πραγματικά ε, ε, παίρνουν κάθε μέρα εκεί στις αγροτικές ε, περιοχές, την καθημερινότητά τους εκεί. Και νομίζω πως σήμερα θα ακούσουμε μία σειρά από πτυχέ σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Εγώ για παράδειγμα έκανα κάποιες σκέψεις σχετικά, δηλαδή τι συμβαίνει όταν το επάγγελμα και η η παράδοση που ακολουθεί ε, κανείς και ο τρόπος ε, ζωής του ε, είναι πολύ στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Για παράδειγμα κάποιος ο οποίος ζει σε ένα αγρόκτημα και φροντίζει και την οικογένεια, φροντίζει και τους γονείς, όλα αυτά αποτελούν κοινά στοιχεία της ζωής στην αγροτική περιοχή. Αυτό είναι ένα μοντέλο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η αγροτική περιοχή όπου η γυναίκα εργάζεται σε ένα σημείο αλλά ε, ζει σε ένα άλλο και ε, αντιμετωπίζει για ε, παράδειγμα προβλήματα μετακίνησης στον τόπο εργασίας και εκεί τίθεται και ερωτήματα ως προς το πώς θα φροντίσει για παράδειγμα για τη φροντίδα των παιδιών, για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, τη διαχείριση της οικογένειας, του νοικοκυριού δηλαδή και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το επάγγελμα και το σημείο διαβίωσης μπορούν να βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους ή να είναι ε, πολύ μακριά μεταξύ τους. Επίσης, το ζήτημα γενικά της κινητικότητας είναι ε, ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αγροτική περιοχή. Επίσης, ένα ακόμα ζήτημα είναι η διαχείριση ε, των καθημερινών δραστηριοτήτων. Πώς μπορεί δηλαδή μια γυναίκα να διαχειριστεί καλύτερα τον χρόνο της στην αγροτική περιοχή, ούτως ώστε να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις. Γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές οι γυναίκες και μάλιστα είναι οι πρώτες οι οποίες εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές όταν η, η κοινωνική δομή σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ εύθραυστη αν θέλετε ή όχι πολύ ισχυρή. Είναι δηλαδή ένα ε, είδος ε, δίκτυ η εγκατάλειψη των ε, αγροτικών περιοχών από τις γυναίκες. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου σχεδόν δεν υπάρχουν πλέον γυναίκες οι οποίες μένουν εκεί και βέβαια αυτό αποτελεί μια πρόκληση τόσο σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής όσο και σε επίπεδο χάρη ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γενικότερο επίπεδο. Άρα λοιπόν χαίρομαι για αυτούς τους λόγους που θα συζητήσουμε για αυτό το σήμερα και ευχαριστώ για μία ακόμα φορά τη συνάδελφα συνάδελφο που πρότεινε τη διοργάνωση αυτού του workshop. Ε, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Νοίσιλ. την ευχαριστώ για τα θετικά της ε, λόγια και να περάσουμε στην ε, πρώτη μας καλεσμένη, την καθηγήτρια Ραμόνα Φράνιτς, που είναι καθηγήτρια πολιτικής και εργοδικής οικονομίας ε, στην, ε, στο Πανεπιστήμιο του Σάγκρεπ στην Κροατία και έχει εξειδικευτεί σε μία σειρά αποζητήματα μεταξύ άλλων στην ε, αξιολόγηση της αγροτικής ανάπτυξης αγροτικές περιοχές τον αντίκτυπο των αγροτικών πολιτικών στην αγροτική οικονομία και στις υπαίθριες περιοχές ε, στην ε, ανάλυση της, ε, του ζητήματος της πτυχής της όντας μεταξύ των δύο φύλων, μεταξύ άλλων και στις αγροτικές περιοχές και την ενσωμάτωση αυτού του ζητήματος στις σχετικές αγροτικές πολιτικές, ειδικότερα στην Κροατία αλλά και στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Οπότε να δώσω κατευθείαν το λόγο στην καθηγήτρια Φράνης. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια στην εισαγωγή σας. Ελπίζω να καταφέρω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτό το workshop που οργανώνεται και να σας μεταφέρω κάποιες από τις εμπειρίες μου από την Κροατία. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις Ανατολικής Ευρώπης. θα σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα μετά από μια ανάλυση της βιβλιογραφίας για τα θέματα αυτά. Ας, ακούσουμε, ας ξαναδούμε ορισμένες από τις πληροφορίες υποβάθρου, τις οποίες φαντάζομαι πολλοί από εσάς γνωρίζετε. Ανέλεσα μεγάλο αριθμό ε, επιστημονικών άρθρων και στοιχείων όσον αφορά τον ρόλο των γυναικών στην αγροτική οικονομία και την οικονομία γενικότερα, είναι ξεκάθαρο ότι οι γυναίκες έχουν ε, πρωταγωνιστικό ρόλο και κύριο ε, ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας και την ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές. Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμάται ότι οι γυναίκες ευθύνονται για την παραγωγή του ίμιση των τροφίμων στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν λοιμό στον κόσμο, 7 στους 10 είναι γυναίκες. Το στοιχείο αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες παράγουν ε, τρόφιμα ε, σε μεγάλο βαθμό έχουν στην κατοχή τους το λιγότερο από το 15% της γης παγκοσμίω και αν κοιτάξουμε τον, τις ανεπτυγμένες χώρες το λιγότερο από το 2% της ε, ιδιοκτησίας ανήκει σε γυναίκες. Βέβαια υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα αλλά κατά βάση τα προβλήματα είναι τα ίδια αυτό που διαφέρει είναι η έντασή τους. Κατά συμπέρασμα, υφίστανται ακόμα διακρίσεις οι γυναίκες, δεν έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου οι γυναίκες να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Χρειάζεται λοιπόν μια στοχευμένη πολιτική για να εφαρμοστεί στην πράξη η ισότητα των δύο φύλων. Ποιοι ήταν οι στόχοι μας ε, σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Θέλαμε να καταγράψουμε συνοπτικά, συγκεντρωτικά την κατάσταση των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη, τον, την θέση τους στην αγορά εργασίας, το ρόλο τους όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων, τον, την θέση τους στην αγορά τροφίμων, τη σημασία που έχει ο ρόλο τους, τους στην βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και επίσης το ρόλο που διαδραματίζουν σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως για παράδειγμα την διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτισμικής ε, παράδοσης καθώς επίσης να εξετάσουμε κατά πόσον οι γυναίκες ε, και πώς οι γυναίκες συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων και στην χάραξη πολιτικών. Το επαναλαμβάνω. Οι γυναίκες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν για να θρέψουν την οικογένειά τους και για, να, για την πρόοδο, για την ευημερία της κοινωνίας τους. με τη δουλειά τους οι γυναίκες δίνουν τροφή ξεκινώντας από τις οικογένειάς τους σε ολόκληρη την κοινότητά τους. Το 2, το, το, το, το, 2 τρίτα αυτής της εργασίας γίνεται από γυναίκες, αλλά το εισόδημα τους ανέρχεται στο 10% του εισόδηματος παγκοσμίως. Οι οικονομικέ ανισότητε λοιπόν είναι τεράστιε και γίνονται ακόμα πιο εμφανεί αν κοιτάξουμε και το ζήτημα τη ιδιοκτησία. Αυτό που σα έλεγα πριν, ότι το 2% ανήκει στι γυναίκε. Επομένω, το θέμα τη ανισότητα των δύο φύλων δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα που αφορά τι γυναίκε. Είναι και ένα οικονομικό πρόβλημα για τι αγροτικέ περιοχέ, το οποίο μετά έχει επιπτώσει στον τομέα τη επιστημιστική ασφάλεια και τη ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών. ο ρόλος του κάθε φίλου ε, όσον αφορά τον καταμερισμό εργασίας έχει βαθιές ρίζες. Ίσως κάποτε να ήταν δικαιολογημένη αυτή η, αυτή η διαφορετική ρόλη των δύο φύλων, αλλά ε, είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα προβλήματα τα οποία συζητήσαμε μέχρι τώρα και συζητούμε θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι ρόλοι των δύο φίλων οι παραδοσιακοί έχουν ξεπεραστεί. Αναφερόμαστε συχνά με τον αγγλικό όρο gender mainstreaming στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών. Και αυτή θα πρέπει να είναι πολιτική ε, που θα ακολουθήσουμε για την καταπολέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εξετάζονται στην 21 των 28 κρατών μελών, πάνω από το 50% είναι γυναίκες φυσικά του πληθυσμού, όμως αν κοιτάξουμε τον ε, οικονομικά ενεργό πληθυσμό, το 46% είναι γυναίκες. Ήδη το πρώτο σημάδι ότι εδώ υπάρχει ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αν κοιτάξουμε επίσης τα στατιστικά στοιχεία της ανεργίας, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες συχνά εργάζονται σε ε, δουλειές με μικρότερο βαθμό, με λιγότερες αρμοδιότητες, με λιγότερες ευθύνες και συχνά χαμηλότερα αμοιβόμενες. Στην Ιταλία, στην Ελλάδα, Ουγγαρία η κατάσταση είναι χειρότερη. Τα στοιχεία για το 2013 μας δείχνουν το 16,6% του πληθυσμού στα 28 κράτη-μέλη βρισκόταν στο όριο της φτώχειας. Και πάλι οι γυναίκες είναι η πλέον ευάλωτη ομάδα να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Με την αύξηση λοιπόν της απασχόλησης θα μειωθεί η φτώχεια θα βελτιωθεί και η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση των μελών της κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα εξετάσαμε τον ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στην παραγωγή τροφίμων. Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές παράγουν πάνω από το μισό των τροφίμων. Σε, αν κοιτάξουμε τις αναπτυσσόμενες περιοχές, ε, αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο 80% ή και περισσότερο. 80%. Ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής δεν καταγράφεται. Για παράδειγμα εκείνοι που έχουν ένα, ένα περιβόλι. Σε αυτά τα περιβόλια συνήθως δουλεύουν γυναίκες. Αυτό το διαπιστώνουμε στην Κροατία και διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτού του τύπου την μη καταγραφόμενη αγροτική παραγωγή και λείπουν τα στατιστικά στοιχεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσαν να μας κάνουν να καταλάβουμε εάν υπάρχει υπάρξει πρόοδος στον τομέα της συμμετοχής των γυναικών στην παραγωγή την αγροτική. Έχω ένα παράδειγμα ε, που αφορά την Ισπανία. Στην Ισπανία διαπιστώνουμε ότι ήταν πάντοτε ευθύνη των γυναικών να φροντίζουν ε, για να έχει φαγητό η οικογένεια. Αλλά κανείς δεν το θεωρεί αυτό οικονομική δραστηριότητα. Το θεωρεί ε, κανείς ε, φροντίδα της οικογένειάς του. Στη Ρουμανία διαπιστώνουμε μεγάλη ε, διαφορά στο εισόδημα ανδρών και γυναικών. Μεγάλο χάσμα. Συχνά ε, οι οικιακές εργασίες δεν αναγνωρίζονται. Δεν αμείβονται και δεν ε, εμφανίζονται και στα στατιστικά στοιχεία. Και γι' αυτό οι γυναίκες ε, κινδυνεύουν περισσότερο από τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Για να μην σα κουράζω με τις διαφάνειες μου, σα έχω και ορισμένε φωτογραφίες. Η κυρία που βλέπετε στην οθόνη σας είναι από την Κροατία, είναι αγρότησα, δεν είναι και τόσο νεαρή ηλικία όπως βλέπετε, αλλά είναι ιδιαίτερα ε, δραστήρια. Δεν θα καταμετρούσε κανείς ε, στον ε, οικονομικά ενεργό πληθυσμό, αλλά επί της ουσίας είναι εξαιρετικά δραστήρια, εκείνη φέρνει το φαγητό στην οικογένειά της και με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει και στη σταθερότητα της κοινωνίας, της κοινότητάς της. Αναφέρθηκα λοιπόν στη σημασία του ρόλου των γυναικών στην αγροτική οικονομία. Όσον αφορά τώρα τις αναπτυγμένες χώρες, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες έχουν σημαντικό ρόλο και στην ε, οικονομία των ε, τροφίμων. Αγοράζουν το 81% ε, των αγορών γίνεται από γυναίκες και το 81% συνολικά το προϊόντο γίνεται από γυναίκες και το 82% όσον αφορά το τρόφιμα. Ε, βεβαίως αυτά είναι συνολικά συγκεντρωτικά στοιχεία αλλά δείχνουν κάτι. Οι γυναίκες είναι εκείνες που προκαλούν τις αλλαγές στην οτροπία των κατανολωτών. Εκείνες προσέχουν, για παράδειγμα, για την ασφάλεια των τροφίμων. Εκείνες φροντίζουν τα τρόφιμα να είναι υγιεινά. Εκείνες φροντίζουν ακόμα και τα τρόφιμα που αγοράζουν να είναι όμορφα. Διαμορφώνουν έτσι λοιπόν την αγορά των τροφίμων. Και έρχομαι τώρα στο ζήτημα της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών. Στην Κροατία πρόσφατα διεξήγαμε μια έρευνα με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Εξετάσαμε τις απόψεις των ε, γυναικών και των ανδρών όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Ορισμένοι, οι, οι άντρε, νομίζουν ότι είναι απλώ οικονομικό το θέμα. Το βλέπουν ω επιχείρηση. Οι γυναίκε έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στο να, στη διατήρηση του τρόπου ζωή του χωριού, την δυνατότητα να ε, φροντίζει κανεί για την οικογένειά του, να φέρνει το φαγητό στην οικογένειά του. Δηλαδή έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα άλλο παράδειγμα από την Πορτογαλία, όπου οι γυναίκες συνεισέφεραν ε, πολύ στην ανάπτυξη του τουρισμού και την αναζωγόνηση των αγροτικών περιοχών μέσω του ε, τουρισμού. Άλλη μια φωτογραφία. Από την Κροατία είναι η κυρία που βλέπετε, αλλά και από την Πορτογαλία θα μπορούσε να είναι. Θέλω να σας ζητήσω στο τέλος της παρουσίασής μου, αν είναι κάτι να θυμάστε, να είναι αυτές οι φωτογραφίες. Κρατάει στα χέρια της ένα ε, πανέρι με σταφύλια. Σας μίλησα για τη σημασία του ρόλου του γυναικών και για την παραγωγή και για την κατανάλωση τροφίμων. Έχουν και έναν ακόμα ενδιαφέροντα ρόλο. Τη διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης. Σε όλες τις μελέτες που εξέτασα, δίνεται έμφαση στο ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στην οικογένειά τους, και τις διαφορετικής νοοτροπίας που έχουν ε, και στο σπίτι αλλά και στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για τα συναισθήματα του συνανθρώπου τους. Ένα παράδειγμα από την Ελλάδα. Μια μελέτη λοιπόν από την Ελλάδα μας δείχνει ότι η δημιουργία μικρών επιχειρήσεων ε, ιδιοκτησίας γυναικών, συνεισέφερε στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων με παραδοσιακούς τρόπους και με αυτόν τον τρόπο βοηθήθηκε και η διατήρηση της παραδοσιακής ε, καλλιέργειας. Πέρα από τα οικονομικά ωφέλη. μια άλλη μελέτη από την Κροατία. Εδώ πήγαν ένα βήμα, παραπέρα οι γυναίκε για την προστασία τη πολιτιστική του παράδοση. Φαντάζομαι θα συμβαίνει και σε άλλε χώρε. Σα φέρω ένα παράδειγμα από την Κροατία, γιατί είναι η χώρα μου και την ξέρω καλύτερα. οι γυναίκε εκεί έχουν συστήσει μη κυβερνητικέ οργανώσει, σωματεία ή και ανεπίσημε ομάδε με τις οποίες οργανώνουν εκδηλώσεις για να μοιραστούν τις παραδόσεις του χωριού τους και να φροντίσουν να μην χαθούν αυτές οι παραδόσεις. Πολύ συχνά έχουμε τέτοια ε, εκδηλώσεις στα χωριά της Κροατίας. Ορίστε ένα παράδειγμα. Η κυρία στα αριστερά της φωτογραφίας είναι η ίδια κυρία που σας έδειξα προηγουμένως στο θερμοκήπιο ε, που καλλιεργεί ε, τις ντομάτες. Εδώ τη δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσει για τις δραστηριότητε τη σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Κάπω έτσι βλέπαμε τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία, στα Βαλκάνια, στην Κροατία. Έραβαν, ε, καλλιεργούσαν, φρόντιζαν τα παιδιά, κοινωνικές ε, πιέσεις, ότι περιμένει κανείς ε, στο χωριό η γυναίκα να έχει φροντίσει το περιβόλι να είναι. Σιγά σιγά όμως αλλάζουν οι νοοτροπίες. Σιγά σιγά βλέπουμε, ωστόσο μάλλον συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι παρά την συνεισφορά τη σημαντική των ε, γυναικών στην αγροτική οικονομία, η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων δεν είναι η επιθυμητή, είναι μικρή. Και δυστυχώ δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξη για το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα εδώ. Το παράδειγμα από την Πολωνία έχει ενδιαφέρον. Συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η φροντίδα των παιδιών ή άλλων ανθρώπων θεωρείται γυναικεία δουλειά. με τέτοιου τύπου δραστηριότητε είναι γνωστές, για τέτοιου τύπου δραστηριότητε είναι γνωστέ οι γυναίκε στι κοινωνίε του, όχι τόσο για αυτό που κάνουν επαγγελματικά. Παρά το γεγονό ότι μελέτε, για παράδειγμα, από τη Σλοβακία μα έχουν δείξει ότι οι γυναίκε μπορούν να είναι πιο επιτυχημένε επαγγελματικά ακριβώ επειδή ξέρουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ή να του ενδιαφέρουν τα προβλήματα των άλλων. Έχουν τη δυνατότητα να ε, λειτουργήσουν καλύτερα σε μικρέ ομάδε ή σε ε, χώρου εργασία με έλλειψη πόρων. έχουν για παράδειγμα την εμπειρία να προσφέρουν στην κοινωνία ε, και έρχομαι στα μέτρα τα νομοθετικά που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 25 χρόνια σε όλες τις, τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένες και τις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, έχει εισαχθεί μια διάσταση φύλου. Αυτό εκφράζεται με συγκεκριμένες νομικές προβλέψεις και συγκεκριμένα εργαλεία για την βελτίωση των συνθήκων των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, την συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. Το ζήτημα βέβαια πάντα είναι κατά πόσον αυτή η νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά και αποτελεσματικά. Και επίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για να μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώ ποιο είναι ο ρόλο των γυναικών. Στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξη τονίζεται η σημασία του ρόλου των γυναικών. Και ορισμένες φορές τους δίνονται και κάποια ιδιαίτερα πλέον εκτίματα, κάποιες ιδιαίτερες επιδόματα ή επιδοτήσεις βοήθεια. Αλλά όχι αρκετά και το γιατί φαίνεται από τις παρατηρήσεις που έκανα στην αρχή της παρουσίασής μου. Συχνά για να λάβει κανείς οικονομική βοήθεια, για παράδειγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοντήλια, πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης μιας εκμετάλλευσης γεωργικής. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στις αγροτικές περιοχές. Στην Ιταλία, οι γυναίκες απολαμβάνουν κάποια προνόμια στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την, για την πρόθεση της επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν ειδικά μέτρα για την πρόθεση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μια μελέτη στη Σλοβενία μας έδειξε ότι το σχέδιο ευρωτικής ανάπτυξης που έχει κατακτήσει αυτή η χώρα και επίσης οι πόροι που δόθηκαν για την αγροτική ανάπτυξη στη χώρα αυτή βελτίωσαν σημαντικά την ε, υποδομή και τις εκμεταλλεύσεις, αλλά δεν βελτιώθηκε η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων. Συμπερασματικά, οι γυναίκες δεν έχουν κατακτήσει ακόμα την ισότιμη θέση που τους αξίζει όσον αφορά την αμοιβή και τις θέσεις εργασίας. Πολύ συχνά η συνεισφορά τους παραμένει αφέατη, επομένω πρέπει να κινητοποιηθούμε. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι τα εμπόδια που σταματούν τις γυναίκες από το να συμμετέχουν ε, ισότιμα στα κοινά και στο τοπικό και ε, στο περιφερειακό και τα λοιπά επίπεδα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Και μιας και προσωπικά ε, εργάζομαι στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θα μπορούσα παρά να αναφερθώ στη σημασία που έχει η ευαισθητοποίηση, η χρήση του εκπαιδευτικού συστήματος να δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες να γνωρίζουν πώς να ε, εξεύρουν πόρους, δάνεια επιδοτήσεις κτλ. Αλλά η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, η εκπαίδευση των γυναικών βεβαίως πρέπει να βελτιωθεί, αλλά αφορά επίσης και τους άντρες που θα πρέπει να εκπαιδεύονται στο ζήτημα της ισότητας. Υπάρχουν θετικές εξέλιξεις, θετικές τάσεις τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Τουλάχιστον σήμερα ε, οι δείκτες και τα κριτήρια και η ανάλυση που σας παρουσίασα είναι ξεκάθαρες, ξεκάθαροι και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και ακόμα περισσότερο στις αγροτικές κοινωνίες. Κλείνω με ορισμένες συγκεκριμένες συστάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να διοργανώνει τέτοιου τύπου συναντήσεις όπως η σημερινή. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε και περισσότερους μετέχοντες σε τέτοιου τύπου συναντήσεις. Είναι σημαντική, όπως σας είπα, η ευαισθητοποίηση του σκηνής γνώμης και η διαρκής εκπαίδευσή της. Αυτό είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση κάθε κοινωνικού προβλήματος, όχι μόνο της ισότητας των δύο φύλων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω έχει στη διάθεσή του πολλές δυνατότητες, πολλά εργαλεία. Πρέπει να εκτιμάται δεόντως η συνεισφορά των γυναικών, είτε αυτές εργάζονται σε μια επιχείρηση, σε ένα γραφείο, είτε σε μια οικογενειακή αγροτική ε, ε μονάδα. Τα στατιστικά στοιχεία που έχει στα διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιωθούν. Οι βάσεις δεδομένων πρέπει να βελτιωθούν. Γιατί ένα μεγάλο μέρος της ε, εργασίας των γυναικών ε, παραμένει στην αφάνεια, δεν, δεν καταγράφεται. Τώρα όσον αφορά τα, το, τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόθεση της γυναικείας επιχειρηματικότητας Και άρα θα πρέπει να, έχουμε, να είμαστε πιο ανοιχτοί στο να ακούσουμε τις δικές τους ιδέες, τις δικές τους προσεγγίσεις. και στο τοπικό και στο εθνικό επίπεδο είναι καλύτερα να προωθήσουμε συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένους στόχους που προωθούν την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών Οι πολιτικές μας δεν θα πρέπει να επιδιώκουν μόνο την ε, εξάλληψη των διακρίσεων κατά των γυναικών ή την ισότητα των δύο φύλων στο επίπεδο της διοίκησης ή του κράτους. Το ζήτημα είναι επίσης κοινωνικό, έχει επίσης ε, σημασία ε, να θεωρείται συμπληρωματική η συνεισφορά των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία. Μόνο αυτό μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία να πάει πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την καθηγήτρια Φράνιτς για αυτή την παρουσίαση. Θα δώσω τώρα το λόγο στην δεύτερη εμπειρογνωμονά μας, την κυρία Τζάνετ Ντουάρ, που έχει ε, ένα μάστερ σε βιολογία και ένα διδακτορικό στην αγροτική οικονομία και είναι ε, καθηγήτρια αγροτικής ε, πολιτικής του Ιδρύματος Ερευνούς για τις Αγροτικές περιοχέ και τις ε, κοινότητε του Πανεπιστημίου του Gloucestershire στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ιδιαίτερη εμπειρία η κυρία Ντουάρ σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των γεωργικών πολιτικών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ακολουθώντας δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά αυτή την αξιολόγηση, οπότε θα της δώσω απευθείας το λόγο. Κυρία Ντουάρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλους που μου δίνετε. Ε, μου δώσατε την ε, δυνατότητα να έρθω σήμερα εδώ. Όπως ε, είπε η Πρόεδρος, έχω κάνει για σειρά ετών έρευνα σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική και την ανάπτυξη της υπέτρου, αλλά δεν έχω εργαστεί ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα ε, των, ε, της, ε, σε των φύλων και γι' αυτό αποτέλεσε για μένα κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Μια πρόκληση δηλαδή προκειμένου να εξετάσω λίγο καλύτερα τη χρηματοδότηση κοινή γεωργική πολιτική σε σχέση με το ρόλο των γυναικών στο πλαίσιο της αγροτική δηλαδή ανάπτυξη και τη και τη ανάπτυξη των υπεύθυνων περιοχών. Άρα μου ζητήθηκε λοιπόν να εξετάσω το πώ η χρηματοδότηση των πολιτικών τη κοινή γεωργική ε, πολιτική επηρεάζει δηλαδή τον ρόλο των γυναικών ε, στην αγροτική οικονομία και στην ανάπτυξη των υπεύθυνων περιοχών. Ε, μου ζητήθηκε το Σεπτέμβριο να διεξάγω αυτή τη μελέτη, οπότε αυτή έγινε στο γραφείο μου, δηλαδή εξετάζοντα τη σχετική βιβλιογραφία στις ε, διάφορες δηλαδή δημοσίευσεις της διάστασης πολιτικής και στα κλαδικά ε, περιοδικά. Επίσης ε, προέβησε μια ανάλυση των δεδομένων που διατίθεται από την ίδια την Επιτροπή και την Eurostat σε ό,τι αφορά τις πτυχές ακριβώς ε, της ε, εκπροσώπησης ε, των φίλων στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής και η ανάλυση αυτή των δεδομένων διεξήχθη προκειμένου να διαπιστώσουμε το αν υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά την απορρόφηση της χρηματοδότησης ε, δηλαδή διαφορέ ανάμεσα σε άντρε και γυναίκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Νίκ Λούι, ο οποίο ε, ήταν όμως για τη διαχείριση των δεδομένων, αλλά να ευχαριστήσω και μια σειρά από άλλε γυναίκε ακαδημαϊκούς από άλλα σημεία τη Ευρώπη που με βοήθησαν πάρα πολύ να ε, βρω την κατάλληλη βιβλιογραφία και με βοήθησαν στο να εστιάσω λίγο καλύτερα το έργο που έκανα. Από την εξέταση λοιπόν τη βιβλιογραφία, στην οποία προέβη, και συμφωνώντας με τα όσα ε, είπε η προηγούμενη, ε, η προηγούμενη ομιλήτρια, η καθηγήτρια Φράνης λοιπόν, προέκυψε ότι στις καλλιέργειες ένα σημαντικό κομμάτι του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες, αλλά το μερίδιό τους ε, ως ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων, δηλαδή από νομικής άποψης, να έχουν ή την διαχείριση των πόρων της εκμετάλλευσης ή να έχουν την νομική κατοχή, είναι πολύ χαμηλότερο το λόγο μερίδιό. Ε, παρόλα αυτά ε, πολλές μελέτες δείχνουν ότι είναι αποφασιστικός ο ρόλος που παίζουν οι γυναίκες σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις ε, καθώς εξασφαλίζουν το να λειτουργεί εύρυθμα αυτή η ομάδα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της εκμετάλλευσης, δηλαδή η οικογένεια. Και υπάρχουν διάφορες μελέτες που εξετάζουν το ρόλο της αγροτικής οικογένειας και της γυναίκας μέσα σε αυτήν σε διάφορες χώρες και παρότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των λόγων χωρών υπάρχουν, διακρίνουμε Διαφορέ ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Αν λοιπόν κάνουμε μια γενίκευση για ε, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπιστώσουμε ότι ο ρόλος της γυναίκας, είναι πολύ σημαντικός τόσο σε ό,τι αφορά τις, ε, τις υπηρεσίες, συνοδευτικές ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη λογιστική, σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση των νεαρότερων ζώων. Έχουμε για παράδειγμα ε, περισσότερη εκπροσώπηση των γενικών στον κλάδο της εκτινοτροφίας από τις θαλωτρές καλλιέργειες και ταυτόχρονα είναι οι οι γυναίκες οι οποίοι εξετάζουν ε, και αναζητούν και άλλους πόρους εισοδήματος από διαφοροποιημένες δηλαδή επιχειρήσεις για παράδειγμα από από από ε, τον τουρισμό και ούτω καθεξής προκειμένου να εξασφαλίσουν πληρωματικό συνόδημα, εισόδημα. Ε, και γι' αυτό ακριβώς έχουν συμμετάσχει πιο ενεργά οι γυναίκες στο πρόγραμμα Leader, το κοινωτικό πρόγραμμα Leader. Εάν ε, εξετάσουμε λοιπόν τώρα το ζήτημα από αναλυτική άποψη, θα δούμε πως ε, τα στοιχεία, τα ακαδημαϊκά στοιχεία, ε, μας δείχνουν ότι καθιστούν πιο ανθεκτικές τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις οι γυναίκες γιατί είναι πιο ευέλικτες και προσπαθούν να εξετάσουν και να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους ε, πόρους που μπορεί να έχει η οικογένεια προκειμένου να είναι και πιο ανθεκτική στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Ταυτόχρονα αυτό που βλέπουμε επίσης να αποτελεί κοινή ε, θέση είναι ε, στη βιβλιογραφία ότι η αναγνώριση αυτή όμως του, του, του ρόλου των γυναικών δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο η αναγνώριση του ρόλου των ανδρών. Και ε, σημειώνεται κάποια πρόοδος και αν έχετε ε, λίγο χρόνο και εξετάσετε ε, την έκθεσή μου θα δείτε το, τις παραπομπές που έχω εκεί σε διάφορες δηλαδή έρευνες που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε ό,τι αφορά γενική νομοθεσία και γενικές πρωτοβουλίες αυτές ε, λαμβάνουν χώρα ε, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα έδος υποστρώματος για την υποστήριξη του ρόλου των γυναικών σε όλους τους τομείς. Αλλά από εκεί και μετά ε, συνδυάζεται αυτή η γενική προσέγγιση με μια ιδιαίτερη έμφαση για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα της ε, και αυτά που ανέφερε η καθήτρια κυρία Φράνης, δηλαδή τρόπους με τους οποίους μπορούμε να καταστήσουμε ευκολότερη την πληρέστερη συμμετοχή των γυναικών με αυτού τους ρόλους. Εδώ η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία είναι παραδείγματα που αναφέρω εδώ και μας δείχνουν διαφορετικά παραδείγματα ε, συστημάτων ή προσεγγίσεων τα οποία επιτρέπουν στις γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο, να είναι πιο ε, να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να παίξουν πιο ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά ε, την επίδραση που μπορούν να έχουν στις αλλαγές στο επίπεδο δηλαδή την, της εκπροσώπησης των δύο φίλων στο κοινωνικό τομέα. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια δέσμευση στο επίπεδο της πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής πολιτικής, σε ό,τι αφορά το mainstreaming, δηλαδή την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινωτικές πολιτικές, αλλά διαπιστώνεται ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η διάσταση στο επίπεδο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η, η κοινή γεωργική πολιτική δεν ε, δεν δίνει την έμφαση αυτήν, δηλαδή έχει σχεδιαστεί με τρόπο ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα ακριβώς ε, ε, της, των διαφορών μεταξύ των δύο φυλών και ακριβώς επειδή είναι ουδέτερη απέναντι σε αυτά τα ζητήματα η βιστάμενη πολιτική δεν μπορεί να επιφέρει και αλλαγές. Υπάρχουν κάποιες μικρής κλίμακας στοχευμένες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τέτοιου είδου μικρέ πρωτοβουλίε δεν μπορούν να επιφέρουν μια γενικότερη αλλαγή. Άρα, διαβάζοντα αυτέ τι αναφορέ και αυτά τα συμπεράσματα των μελετητών αυτών των ζητημάτων εδώ και χρόνια, ε, σκέφτηκα να εξετάσω τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μα ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και να, δω, ε, και να δούμε κατά πόσο πράγματι αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν αυτά τα συμπεράσματα των μελετητών. Ε, εν είδη εισαγωγή λοιπόν σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μα, Εδώ αναφέρομαι σε δεδομένα από την Eurostat σε ό,τι αφορά την διάθρωση των εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξέταση του ποιο είναι ο κύριο αρμόδιος, ο κύριο διαχειριστή ε, τη λόγω εκμεταλλεύση. Οπότε αριστερά ε, στο γράφημα βλέπουμε ε, αυτή την, ε, την, την διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλλα για το έτος 2010, γιατί έχουμε τα πληρέστερα δεδομένα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κοντιλίων από αυτές τις εκμεταλλεύσεις και βλέπουμε λοιπόν ότι στο σύνολό τους οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις ανήκουν σε άνδρες. Ε, είναι μικρότερο το μερίδιο των ε, γυναικών και έχουμε και ένα αυξανόμενο μερίδιο σε μια σειρά από κράτη-μέλη ε, επιχειρησιακές ιδιοκτησίες, δηλαδή κάποιες ε, κάποιο είδους ε, εκμετάλλευση δηλαδή όπου έχουμε επιχειρηματικού χαρακτήρα Για παράδειγμα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε πάντοτε μεγάλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, στη Γαλλία μιλάμε απλά για επιχειρηματικού χαρακτήρα εκμεταλλεύσεις οικογενειακές. Οπότε δεν σημαίνει αυτομάτως όταν βλέπουμε corporate, όταν βλέπουμε δηλαδή ότι έχουμε επιχείρηση ως ιδιοκτήτη ότι μιλάμε για μέγαλο επιχειρήσεις. Αλλά βλέπουμε λοιπόν εδώ στο, στο γράφημα ε, της, ε, ε και βέβαια εδώ η κλίμακα είναι λογαριθμική. Ε, στα δεξιά και βέβαια και αυτό γιατί θα βρίσκονταν πολύ πιο ε, ψηλά σε αυτή την κλίμακα οι ε, εκμεταλλεύσεις. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν το μέσο όρο και διαπιστώνουμε ότι οι εκμεταλλεύσεις ή ε, το μέγεθο των εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε γυναίκες ε, είναι, ε, βρίσκεται στο ίμιση αυτών που ανήκουν στους άντρες και βέβαια είναι πολύ μικρότερο το μέγεθος σε σύγκριση με αυτό που, των εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε επιχειρήσει. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό έχει και σημασία σε επίπεδο πολιτική. Αν δούμε τον πρώτο πυλώνα της κοινή γεωργική πολιτική μετά από 20 χρόνια μεταρρυθμίσεων βρισκόμαστε σήμερα σε μια φάση όπου η μεγαλύτερη ε, καταβολή γίνεται ε, με βάση το εκτάριο. Και αν ε, αναλογιστούμε το προηγούμενο γράφημα ότι δηλαδή οι εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε γυναίκες είναι γενικότερα μικρότερου μεγέθους, τότε είναι λογικό ότι οι γυναίκες λαμβάνουν και λιγότερες χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του πυλώνα 1 από ό,τι άνδρες ή από ό,τι επιχειρήσεις. Αλλά βέβαια αυτή η ε, ε, διαφορά ε, διαφοροποιείται ανά κράτο μέλο. Δηλαδή σε ορισμένα κράτη-μέλη μπορούμε να μην δούμε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση, αλλά σε γενικέ γραμμέ υπάρχει. Ένα στοιχείο στο οποίο επίσης πρέπει να εστιάσουμε είναι επειδή οι ενισχύσει ορίζονται με διαφορετικό τρόπο έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, σε ορισμένα κράτη-μέλη οι ε, πολύ μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις εξαιρούνται, δεν είναι επιλέξιμες και σε, άλλες, ε, σε άλλα κράτη-μέλη δεν λαμβάνονται υπόψη εκμεταλλεύσεις ε, μερικής, εκμεταλλεύσεις, μερικής απασχόλησης. Οπότε και αυτό επηρεάζει και τον, την εκπροσώπηση των γυναικών. Και βέβαια τίθεται το ερώτημα, αυτό πρόκειται για ένα τους έμεση ε, διακριτική ε, μεταχείριση. Αυτό εξαρτάται από τα κριτήρια που θέτει κανεί. Αν θέλει δηλαδή να συμπεριλαμβάνει τι μεγάλε ε, εκμεταλλεύσει που ανήκουν σε επιχειρήσει και όχι τι πολύ μικρέ, πάνω σε αντικειμενικά κριτήρια. Έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση το γιατί δηλαδή έχουμε τόσο μεγάλο μέρος ε, των χρηματικών ενισχύσεων που πηγαίνουν ακριβώς στις επιχειρήσεις και στις εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε επιχειρήσεις και θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε το κατά πόσο οι στόχοι που έχουν τεθεί αντιστοιχούν στην, ε, στις εξηγήσει που μας δίνονται για αυτήν την εστίαση στις ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ένας από τους στόχους του πυλώνα 1 είναι η υποστήριξη του εισοδήματος. Άρα λοιπόν αντικειμενικά ε, είναι, ε, είναι σωστό να εστιάζουμε κάτι τέτοιο, ε, δηλαδή κάτι που στοχεύει στην, στην ενίσχυση του εισοδήματος σε μεγάλες ε, εκμεταλλεύσεις. Μετά, ε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των, ε, των διών, είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι εκτάσεις στις οποίες διαχειρίζεται κανείς, τόσο περισσότερη χρηματοδότηση χρειάζεται. Αλλά είναι διαφορετικές οι ερμηνείες που μπορούν να δουν εδώ, αναλόγως με το που θα το προσεγγίσει κανείς. Μετά, αν δούμε τον πυλώνα 2, δηλαδή σε ό,τι αφορά την, τις χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, εδώ έχουμε μερικά δεδομένα, όχι πλήρη δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Eurostat, αλλά ε, προ το παρόν τα καλύτερα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μα ήταν το 2010, ε, τα οποία αντιστοιχούν στο περίπου 50% των ε, κοντιλίων και το κυριότερο τμήμα που δεν έχει περιληφθεί υπόψη είναι τα, οι περιοχές of national constraint όπως λέγονται ε, στα αγγλικά, αλλά οι οποίες σε μεγάλο βαθμό της θα λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον πυλώνα 1. Ε, εν πάση περιπτώσει εδώ ε, μπορείτε να δείτε ένα γράφημα, έχετε και τους αριθμούς στην έκθεσή μου. Βλέπουμε λοιπόν το συνολικό δηλαδή των, των, των κατόχων των εκμεταλλεύσεων, δηλαδή αν ανήκουν σε άντρα, σε γυναίκα ή σε επιχείρηση, αριστερά λοιπόν, στην αριστερή πλευρά του γραφήματος βλέπουμε πάλι αυτή την κατανομία ανακάτω μέλους και στη δεξιά πλευρά του γραφήματο βλέπουμε την απορρόφηση ε, των ε, κονδυλίων στο πλαίσιο της, ε, των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Και θα διαπιστώσετε λοιπόν εδώ ότι στις περισσότερες χώρε, η απορρόφηση αυτών των κονδυλίων από τι γυναίκε είναι αναλογικά χαμηλότερη από ό,τι το ποσοστό των γυναικών που είναι κάτω εκμεταλλεύσεων. Άρα λοιπόν Ε, βλέπουμε κάτι το οποίο θα ανέμενε κανείς διαφορετικό, δηλαδή η απορρόφηση να είναι υψηλότερη, ειδικότερα να λάβουμε υπόψη μας ε, την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στις εκμεταλλεύσεις. Ε, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ε, σε σύγκριση με το μερίδιο που καταλαμβάνουν οι ε, επιχειρήσει σε επίπεδο κατόχου της εκμετάλλευσης λαμβάνουν ένα δυσανάλογο υψηλό ποσό, απορροφούν ένα δυσανάλογο υψηλό κοντιλίων αλλά σε ό,τι αφορά ε, τις ε, γυναίκες συγκεκριμένα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σε μια σειρά από χώρες και ε, σε αυτές τις χώρες η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι έχουν, γίνει κάποιες, ε, έχουν ληφθεί ακριβώς κάποια μέτρα, έχουν γίνει κάποιε ε, πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών, οπότε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά ακριβώς τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε το ποια είναι τα πιο δημοφιλή μέτρα. Για παράδειγμα, μία από τις χρηματοδοτήσεις είναι για τον εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και εδώ βλέπουμε τη μεγαλύτερη ανισορροπία ε, ε, ε, μεταξύ δηλαδή των φύλων και της απορρόφησης των κοντιλίων από τις αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις και εδώ δυσανάλογα υψηλό το ποσοστό των επιχειρήσεων και βλέπουμε ότι οι γυναίκες σε γενικές γραμμές είναι πολύ λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στις λόγω χρηματοδοτήσεις για τον εξυγχρονισμό. Τώρα αν δούμε άλλα μέτρα Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση της ε, εκμετάλλευσης, της ε, δημιουργίας προσθέμενης αξίας και της δραστηριοποίηση στον ε, τουρισμό. Οπότε εδώ θα αναμέναμε ότι οι γυναίκες ακριβώς επειδή διαφοροποιούν περισσότερο το εισόδημα της οικογένειας έχουν υψηλότερη εκπροσώπηση και πράγματι αυτό ισχύει, αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνουν στο βαθμό εκπροσώπηση ε, των ανδρών. Βέβαια τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και πάλι τα κράτη-μέλη εκείνα όπου βλέπουμε να έχουν ένα υψηλότερο ποσοστό των γυναικών να εκπροσωπούνται, είναι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία η βιβλιογραφία μα λέει ότι έχουν προωθήσει ιδιαίτερα το ζήτημα τη εξορρόπηση ε, των δύο φύλων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αν η εν λόγω πολιτική ε, επιδιωχθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε αυτό απηχείται και στις, ε, στην απορρόφηση των ε, κοντιλών των προπολογισμών του, για την αγροτική ανάπτυξη. Αν τώρα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τις αιτίε του, γιατί δεν είναι δικαιούχοι, δεν είναι επιλέξιμες οι γυναίκες για αυτές τις ε, χρηματοδοτήσεις, αυτά έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της μη ισορροπημένης εκπροσώπησης των γυναικών. Επειδή δηλαδή οι, σε γενικές γραμμές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε γυναίκες είναι μικρότερης έκτασης, επειδή το επίπεδο κατάρτισης ή εκπαίδευσης των γυναικών είναι σε νητήρες γραμμές χαμηλότερο και επίσης επειδή υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, δηλαδή η εκπαιδευσης των γυναικων ειναι σε γραμμες χαμηλοτερο και επισης επειδη υπαρχει μια διαφορα ηλικία δηλαδη οι αρμοδιοι για τις εκμεταλλεύσεις, οι γυναίκες που είναι αρμόδιοι για εκμεταλλεύσεις σε γενικές γραμμές έχουν μεγαλύτερη ηλικία από ότι οι άνδρες. Και αν εξετάσουμε από αυτό το πρίσμα τις διαφορές θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν, ε, ότι δικαιολογούνται έτσι αυτές οι οι διαφορές. Ε, δηλαδή δεν είναι ότι η ίδια η πολιτική ε, εισάγει ε, δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά στο προφίλ, αν θέλετε, δημιουργούνται αυτές οι διαφορές. αλλά δεν είναι πάντα συνεπής η βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά αυτά τα προβλήματα. Τι μας λένε λοιπόν αυτά τα δεδομένα, ότι σε γενικές γραμμές οι όσοι λαμβάνουν ε, τη, τη χρηματοδότηση αυτό το μέτρο αγροτική αναπτύξης έχουν μικρότερη ηλικία, έχουν περισσότερη κατάρτιση και έχουν μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Και πάλι τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πρόκειται εδώ για μια έμεση δυσμενή διάκριση εις βάρος των γυναικών. θα πρέπει να θέσουμε και πάλι το ερώτημα, αυτές οι αποφάσεις δηλαδή να δίνεται προτεραιότητα στους ε, νεότερους με καλύτερη εκπαίδευση, ε, αγρότε με μεγαλύτερε εκμεταλλεύσεις δικαιολογημένα. Ε, έχει νόημα για να επιτευχθούν οι στόχοι. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει ναι, σε άλλε όμω πάλι όχι. Ε, και ε, αναφέρεται για παράδειγμα ότι θα πρέπει κανείς να έχει τις κατάλληλες, τα, τα κατάλληλα, τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες και ένα αντίστοιχο επιχειρηματικό σχέδιο και μπορεί να ακούγεται αντικειμενικό αυτό θεωρητικά αλλά εάν δεν έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα οι γυναίκε να αποκτήσουν τέτοιου είδου επαγγελματικά προσόντα και αν δεν ε, έχουν ε, τη δυνατότητα να επενδύσουν σε αυτή την ε, επιχειρηματική, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, θα έχουν λιγότερη πρόσβαση στα κονδύλια. Επίση, ε, ε, όποιος θέλει να, συμμετάσχει στη χρηματοδότηση θα πρέπει να ε, ε, βασιστεί και σε πιστώσεις. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες και πάλι θα έχουν λιγότερη πρόσβαση σε πιστώσεις και άρα ε, λιγότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με με, την, με την εμπιστοσύνη που έχουν στον εαυτό τους οι γυναίκες ως ε, ε, διαχειριστές μια τέτοια εκμετάλλευση. Ε, και αυτό βέβαια ισχύει γενικότερα για ε, ε, ομάδες που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό, ότι δεν έχουν δηλαδή τόσο αυτοπεποίθηση. Και βέβαια αυτό μπορεί να βασίζεται και στο γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, που είναι αρμόδιες δηλαδή για την επιλογή, δεν ε, εστιάζουμε μέχρι αλλά θα μπορούσε να αλλάξει αυτό, ε, αυτό ακριβώς εάν οι αρμόδιες αρχές έδειχναν ευαισθησία απέναντι στα ζητήματα, για παράδειγμα του κοινωνικού αποκλεισμού ή τη θέση των γυναικών. Αν παραμείνει ουδέτερη η της θεσης των γυναικων αν παραμεινει ουδετερη η προσεγγιση του, τότε δεν θα αλλάξει ε, κάτι. Ε, Επίση, να πούμε ότι σε σχέση με αυτή την μη ισόρροπη ε, εκπροσώπηση γυναικών ανδρών και σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις θα δούμε πάλι ότι λιγότερο εμφανίζεται στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν λάβει σχετικά μέτρα. Άρα λοιπόν συμπερασματικά ε, τα όσα λαμβάνουμε και από την ε, βιβλιογραφία και από τα δεδομένα ότι είναι ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν προωθεί ε, σοβαρά την ε, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, παρότι δεν κάνει βέβαια, δεν προβαίνει και σε δυσμενέ διακρίσει. Ε, επίσης, εκείνο που είναι ε, ενθαρρυντικό είναι, με βάση δηλαδή τη βιβλιογραφία, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τα μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης, είναι ότι μπορούν πραγματικά να παίξουν σαν αποφασιστικό ρόλο για την ε, περισσότερη, την πιο σοβημένη εκπροσώπηση των γυναικών. Άρα λοιπόν, ε, κατά δική μου άποψη, θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη και το οποίο υφίσταται ε, για να βοηθήσει ακριβώ την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων προκειμένου να επιτευχθούν τα στόχοι των κρατομελών σε περιφερειακό επίπεδο. Άρα λοιπόν, τα εν λόγω κονδύλια θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με τρόπο ούτως ώστε ούτω ώστε να προωθήσουν ακριβώ την καλύτερη ισότητα μεταξύ των φίλων για παράδειγμα με καλύτερη εκπαίδευση, με ε, διοργάνωση εκδηλώσεων σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και προκειμένου να προωθήσουν αυτή την ιδέα ότι δηλαδή είναι δυνατή αλλαγή αν κανεί κινηθεί επικοδομητικά. Και κάτι ακόμα το οποίο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι ότι αν υπάρχει τέτοια βούληση γενικά στο επίπεδο τη πολιτική για το gender mainstream, για την ένταξη δηλαδή τη διάσταση του φίλου στι γενικέ ε, πολιτικέ, τότε γιατί δεν ε, λαμβάνουμε καλύτερα υπόψη υπόψη ε, μας τις οδηγίες που δίνει η Επιτροπή στα κράτη-μέλη ε, στο επίπεδο της εφαρμογή των πολιτικών. Δηλαδή, να γίνεται πολύ πιο ρητή αναφορά και στους δύο πυλώνε τη κοινή ε, γεωργική πολιτική, στα ζητήματα της διάστασης των φύλων. Εγώ συμμετείχα στην ομάδα εκείνη η οποία συμμετείχε στην αξιολόγηση των ενδιάμεσων αξιολογήσεων των ε, προγραμμάτων για την αγροτική αναπτύξη και προσπαθούσαμε να βρούμε εκεί ε, κάποιες λύσεις ότι τι είπαν οι περισσότεροι αξιολογητές σε ό,τι αφορά την ε, διάσταση του φύλου και μας είπαν ότι πολύ λίγα συμβάνουν, δηλαδή δεν λαμβάνει κάτι χώρα σε επίπεδο προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου και βέβαια κάτι τέτοιο να είναι επαρκές θα έπρεπε, να γίνουν πιο πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγα ακόμα λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε θα δώσω το λόγο. Η κυρία Μπεσέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευτυχώς έχουμε ακόμα διερμηνία. Να ευχαριστήσω τις δύο μιλήτριες που μας παρουσίασαν μια εξαιρετική εικόνα από δύο διαφορετικά πρίσματα βέβαια της ε, πραγματικότητας ε, της αγροτικής ζωής. Ε, το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ε, ημέρα, την ε, Διεθνή ημέρα των γυναικών στην αγροτική ζωή, μας δείχνει πόσο σημαντικά είναι όσα έκαναν και πόσο συνεισφέρουν οι γυναίκες και τι ρόλο μπορούν να προάγουν για την προώθηση της ανάπτυξης, την ανάπτυξης με τη γενικότερη έννοια του όρου. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό Αφού καταφέραμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το θεματολόγιο 2030 και τους στόχους ανάπτυξης για το 2030, έχουμε αρχίσει να μιλούμε ε, για το τι ακριβώς ε, μπορούν να συνεισφέρουν οι γυναίκες ε, παγκοσμίω και κυρίως οι γυναίκες αγρότησες. Οι γυναίκες είναι το 50% των χεριών της αγροτικής ε, δύναμης και ε, είναι αυτές οι οποίες ε, χρησιμοποιούν περισσότερο τα χέρια τους, ετοιμάζουν, παρασκευάζουν τροφές και φυσικά όπως και σε πολλούς άλλους τεμές ε, δεν αποτελεί εξαίρεση ανισότητα που εμφανίζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να δούμε γιατί δεν λειτουργούν οι περισσότερες πολιτικές. Αν θέλουμε να υπάρχει συνέπεια στις πολιτικές μας θέλουμε να χρησιμεύουν για το σκοπό που έχουν ε, δημιουργηθεί και αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτές οι πτυχές ε, τις οποίες αναφέρατε και εσείς που σχετίζονται όχι μόνο με τον τρόπο ε, στον οποίο εστιάζουν οι ενισχύσεις ώστε τα διάφορα κριτήρια ανισότητας ε, να οδηγούν τις γυναίκες αγρότησες σε μεγαλύτερες ανισότητες και σε περισσότερες διακρίσεις. Εγώ θα ήθελα να τονίσω, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω, ένα στοιχείο κλειδί για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ελευθερία και τη χειραφόητηση των γυναικών. Είναι ε, η ιδιοκτησία των εκμεταλλεύσεων. Μέχρι τώρα, ε, από όσων ενημερώθηκα, στην Ισπανία και στην βελγική περιοχή της Βαλαιονίας υπάρχει ένα ε, ε, ειδικό καθεστώς συνειδιοκτησίας της ε, εκμετάλλευσης. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε πλήρη νομική ισότητα. Έμεινε απλώ κενό γράμμα η ωραία διάταξη αυτή που υπήρχε και επειδή μέχρι τώρα δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση και επειδή οι γυναίκες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συνειδιοκτησία ε, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι από τις 500.000 ε, υποψήφιες μόνο 136 κατάφεραν να αποκτήσουν συνειδιοκτησία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ε, σημαντικό το στοιχείο αυτό και είναι εξαιρετική ημέρα για να μπορέσουμε να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη, δεδομένου ότι έχουμε και τη Διεθνή ημέρα για τις αγρότησες, να λάβουν υπόψη τους ε, τις συστάσεις αυτές και επίσης ε, να ε, προωθήσουν αυτό το σύστημα κοινή συνειδιοκτησίας όπου να λαμβάνονται τα πάντα αυτομάτως υπόψη λόγω αυτής της συνειδιοκτησίας. Να μην πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε να είναι κάποιος συνειδιοκτήτης, αλλά να υπάρχουν αυτομάτως όλες αυτές οι δυνατότητες και να ενισχύσουμε τα επιχειρηματικά δίκτυα για τις γυναίκες, να υπάρχουν και θέματα κοινωνικής προστισίας, αναγνώρισης ε, του καθεστώτος της συζύγου ως συνειδιοκτήτρια στην εκμετάλλευση, καθώς επίσης ε, και ιδιοκτησία στις υποδομές, στις εγκαταστάσεις και των απαραίτητων για την καθημερινή διαβίωση. Ε, σε μια αγροτική εκμετάλλευση. Αυτό το αίτημα θα το διαβάσω και σε όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής αλλά και άλλων αρμοδίων επιτροπών όπως για παράδειγμα την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την Επιτροπή Γεωργίας. Θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, μια πραγματική ε, ισότητα και να γίνουν πραγματικά ισότητα όλα τα θέματα τα οποία προσπαθούμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Ε, συμμετέχω στην Επιτροπή Μαθημάτων των Γενετών και στην ε, ε, Επιτροπή για τα γεωργικά ζητήματα, οπότε με ενδιαφέρουν πολύ και οι δύο πτυχές. Σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε, σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή και την ενίσχυση ανά εκτάριο, ακούσαμε τα όσα είπατε και ακούσαμε για παράδειγμα ότι τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα παράγονται αν θέλετε από χέρια ανδρών. Ε, οπότε στον δεύτερο πυλώνα είπατε ότι υπάρχει περισσότερη διαφοροποίηση παρότι βέβαια δεν έχουμε ισορροπή εξορροπήση μεταξύ άντρων και γυναικών. Ε, να πούμε ότι εδώ βέβαια μιλάμε για συμπληρωματικό αν θέλετε εισόδημα. Δηλαδή ε, ο πρώτος πυλώνας αφορά εισόδημα ανακτέρω, ο δεύτερος πυλώνας συμπληρωματικό εισόδημα. Οπότε δεν μιλάμε εδώ για υπηρεσίες αν θέλετε οι οποίες έχουν ε, παρασχεθεί, ε, έχουν ε, για δουλειά η οποία αν θέλετε έχει γίνει έργο το οποίο έχει καταβληθεί στον αγροτικό τομέα. Αλλά θα ήθελα να ακούσω για παράδειγμα στο πλαίσιο των συμπληρωματικών αυτών υπηρεσιών για τον τουρισμό ποια είναι τα κονδύλια τα οποία έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο του δεύτερου ε, Γιατί βέβαια η διαφοροποίηση στο αγρόκτημα για παράδειγμα μέσω ακριβώς μια μικρής ε, ξενοδοχειακής μονάδας ας πούμε ενός ε, ξενώνα μέσα στο ίδιο το αγρόκτημα θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον ειδικότερα για τις γυναίκες που αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο οπότε ε, ε, θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω κάτι σε σχέση με αυτό Άλλωστε και στη δική μου περιοχή από την οποία κατάγομαι εγώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ λέει πρώτος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας όμως. Θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα ή στο τέλος. Αφού ακούσουμε τις ομιλωτές. Οπότε καλώς να δώσω το λόγο στους δύο προσκεκλημένες μας. Ή μάλλον θα δώσω το λόγο στην κυρία Πετέν. Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, προσκεκλισμένες μας, τις κυρίες Φράνιτς και του Άιερ. Συνάδελφοι, χαίρομαι που στο τέλος αυτού του εργαστηρίου, επί τη ευκαιρία της ε, Διεθνούς ημέρας ε, των γυναικών στον αγροτικό τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο που ξεκίνησε το εργαστήριο αυτό. Ακούσαμε τα διάφορα στοιχεία που μας είπαν οι ολιμιλήτριες. Είμαι βέβαιη ότι τα βρήκατε πολύ ε, ενδιαφέροντα, όπως τα βρήκα και εγώ, και σίγουρα θα υπάρχουν κίνητρα για να προωθήσουμε το ρόλο των γενικών στις αγροτικές περιοχές. Ε, χαίρομαι επίσης που η Επιτροπή ε, Γυναικών δέχτηκε την πρότασή μου να διοργανώσουμε αυτό το εργαστήριο. Πραγματικά ε, να διατηρηθεί η ζωή στις αγροτικές περιοχές και φυσικά γνωρίζετε ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο. Οι γυναίκες που ζουν στις περιοχές της υπαίθρου παράγουν τρόφιμα, προστατεύουν το περιβάλλον και κρατούν την οικογένεια ενωμένη. Ε, προωθούν την, τον ε, πολιτισμό, την ταυτότητα και τη γλώσσα κάθε έθνους και επομένω χωρί τι γυναίκε τη υπαίθρου δεν θα υπήρχε τοπική κοινωνία. Δυστυχώ ε, ο ρόλο των γυναικών αγροτών δεν αναγνωρίζεται και δεν ε, ε, εκτιμάται επαρκώ. Και αυτό γιατί είναι συνήθως ταπεινές και υπομονητικές, ε, το οποίο ίσως μπορεί να σας κάνει να θεωρήσετε ότι εργάζονται ε, ακάματα όλη την ημέρα. Ε, αλλά ο λόγος είναι κυρίως γιατί δεν αναγνωρίζεται ο ρόλος τους λόγω διακρίσεων και ε, ε, το 80% των γυναικών που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές δεν μπορούν να εξοικονομήσουν καν προς το ζουν. Ορισμένες φορές δεν πληρώνονται για το έργο τους, το αναφέρει η κυρία Φράνιτς άλλωστε, και πολλές από αυτές δεν διαθέτουν καν κοινωνική ασφάλιση ή σύνταξη. Και όταν ε, γεράσουν, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, διότι είτε λαμβάνουν μια πολύ χαμηλή σύνταξη, είτε δεν λαμβάνουν καθόλου σύνταξη. Χαίρομαι που η ε, Επιτροπή μας ε, ενέκρινε την τροπολογία μου για να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να, υποβα... να ε, εισαγάγουν το σύστημα της κατώτατης σύνταξης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολιτικοί συνήθως δεν ενδιαφέρονται για την κατάσταση των γυναικών ε, ε, που εργάζονται στον αγροτικό τομέα και δεν αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους πλήρων. Γι' αυτό ακριβώς ε, ζήτησα να υπάρχει το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις γυναίκες αγρότησες. Την υποστήριξε την ιδέα Επιτροπή μας και ελπίζω στο επόμενο στάδιο να λάβει και την απαραίτητη υποστήριξη. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες αγρότησες και πρέπει να τους προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν και τις θετικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να δημιουργήσουμε ισχυρέ και βιώσιμε αγροτικέ περιοχέ, τι οποίε οι γυναίκε θα διαδραματίζουν κομβικό ρόλο και πρέπει να τι υποστηρίξουμε και να αξιολογούμε το έργο του. Γι' αυτό ακριβώ και γίνεται το σκημερινό εργαστήριο. Δυστυχώ βέβαια είναι περασμένη ώρα, μακάρι να έχει γίνει νωρίτερα γιατί έτσι ε, θα είχαμε περισσότερου ε, βουλευτέ, Ξέρουμε ότι την Πέμπτη το απόγευμα φεύγουν οι ευρωβουλευτέ, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα λάβουν τι πληροφορίε που λάβαμε κι εμεί. Έτσι θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε ε, σε αυτές τις με αυτές τις σκληρά εργαζόμενες γυναίκες. Μπορεί να μην είναι πολύ αλλά έχουν ε, εγγενή σοφία και ένα η αγάπη για τα όσα κάνουν. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τις υποστηρίξουμε και να ε, υποστηρίξουμε τα όσα κάνουν. Ευχαριστώ την κυρία Πετήρα. Α, θα ήθελα να δώσω λόγο τώρα στους προσεκλημένους μας, αλλά θα ήθελα πραγματικά να τους ε, ζητήσω να παρέμβουν μόνο για ένα με δύο λεπτά, γιατί οι διερμηνείς μας θα αποχωρήσουν. Οπότε να ξεκινήσουμε την κυρία Γουάρ. Σας ευχαριστώ. Και πάλι σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή την κουβέντα και να διαπιστώσω ότι το ζήτημα αυτό, τη σημασία του ζητήματος αυτό την αναγνωρίζουν και άλλοι. Και συμφωνούν μαζί μου από αυτό. Επίζω να δοθεί ευρύτερη δημοσιότητα στα αποτελέσματα της μελέτης μου. Μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο για το περιοδικό Agri Europe και σίγουρα με αυτό που άκουσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα προσθέσω και άλλα στοιχεία και ε, οποιοδήποτε έχει κάποιες επαφές με την Επιτροπή Γεωργικής Ανάπτυξης, την Άγκρη, θα μπορούσε να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες. Και εγώ ε, προετοιμάζω ε, μια σχετική μελέτη για εκείνους, θα το κάνω από την πλευρά μου. Κυρία Φράνιτς, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα ακριβώς το ερώτημα, αλλά θα δώσω μια γενική απάντηση. Έχω μπροστά μου έναν πίνακα με αριθμητικά στοιχεία. Διαπιστώνουμε από αυτά ότι οι γυναίκες δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της εστίασης και στον τουριστικό. Ενώ όσον αφορά τα παραγωγή τροφίμων και τη μεταποίηση τροφίμων και εκεί οι γυναίκες στη συμμετοχή τους ξεπερνά το 50%. Οποιοδήποτε πρόγραμμα ενίσχυσης των γυναικών θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα προσαρμοσμένο στο ρόλο που από τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι παίζουν οι γυναίκες. Ε, δεν είχα μια ε, επιστημονικά τυπική μεθοδολογία. Σας έδωσα περισσότερο κάποια παραδείγματα κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Ήθελα περισσότερο να σας μεταδώσω τις εμπειρίες μου από project τα οποία υλοποιήσαμε στην Κροατία. Ένα παράδειγμα. Είχαμε οργανώσει μια ημέρα όπου θα δίδεται ένα βραβείο για τις γυναίκες αγρότησες. Μια κυρία ε, συμμετείχε. Ήταν σύζυγος ενός αγρότη, είχαν έρθει και οι δύο και μου είπε το εξή. Και εγώ ασχολούμαι με την κτηνοτροφία και εγώ ταΐζω τα ζώα που έχουμε, αλλά όταν οι τοπικέ αρχέ οργανώσαν ένα σεμινάριο, προσκάλεσαν τον άντρα μου και εκείνο πήγε και εκείνο θα λάβει τι τελικέ αποφάσει. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Ε, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ να δώσω το λόγο και στην απόσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πριν έρθω εδώ είχα προετοιμάσει κάποια στοιχεία τα οποία ε, πιστεύω ότι έχουν μεγάλη σημασία για, τα, για το θέμα που συζητάμε σήμερα. Στα γρήγορα. Ε, η ισότητα των δύο φύλων έχει ενταχθεί στην υλοποίηση ε, της πολιτικής μας και την παρακολούθηση και της, την αξιολόγηση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία ε, προβλέπουν τις λεγόμενες εκ των προτέρων ερεσιμότητες εξάντε. Ερεσιμότητες δηλαδή εξετάζεται κατά πόσον ο δικαιούχος θα έχει τις διοικητικές υποδομές που χρειάζονται για να υλοποιήσει το έργο, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ισότητα, οι πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων. Μετά, εξασφαλίζεται η συμμετοχή των φορέων για την ισότητα των δύο φύλων. Πιο συγκεκριμένα στα αγροτικά ταμεία, στα ταμεία της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η Γενική Αρχή της Ισότητας των Διοφύλων έχει εξειδικευτεί με θεματικά υποπρογράμματα με συγκεκριμένους στόχους να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Αυτό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά, στο εθνικό επίπεδο, κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τα δικά του κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων κάθε κράτο μέλος, αν μιλάμε για ένα εθνικό πρόγραμμα ή σε μικρότερο επίπεδο, σε χαμηλότερο επίπεδο, οι τοπικές αρχές. Μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα σύστημα συστημα παρακολουθηση με δείκτες, δείκτες μέτρησης της πρόοδου. Από αυτά τα στοιχεία συντάσσονται εκθέσεις ε, οι οποίες θα υποβληθούν το 2017 η πρώτη και το 2019 η δεύτερη. Είναι οι εκθέσεις για την εφαρμογή της ΚΑΠ, ε, της αναθεωρημένης ΚΑΠ. Τότε θα έχουμε τα στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή μας για να δούμε εάν βελτιώθηκε η κατάσταση. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα που ήθελα εγώ να αναδείξω. Με άλλα λόγια, δεν έχω μαζί μου τα στοιχεία ε, που ζητάτε. Ε, μπορούμε ίσως να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας διμερώς για να δούμε ποια στοιχεία θα μπορούσα να σας δώσω. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις ε, και το ότι ήσασταν στη διάθεση σήμερα, σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τις δύο εμπειρογνωμονές μας για το έργο που έκαναν και σίγουρα δεν τελειώνει σήμερα εδώ το έργο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς για την υπομονή που έκαναν για τα 5 παραπάνω λεπτά και η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα είναι το Νοέμβριο σίγουρα 12 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ.